Morning. Buenos días. Buenos días. I have your attention. We should get going. Because we're going to have a busy schedule. Καλημέρα σας, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πρέπει να ξεκινήσουμε και έχουμε και ψηφοφορία κάποια στιγμή αργότερα. Έχουμε τον Έλληνα Υπουργό, οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε με το πρώτο σημείο έγκριση της διατάξη, διατάξεων δεν έχουμε κάποια ε, ένσταση. Έχουμε την αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, ε, στην Ελλάδα και έτσι ανακοινώσουμε τα εξή. PNR στην Ολομέλεια αποφασίστηκε να αναπαιμφθεί δυνάμει του άρθρου 175 το σχέδιο της έκθεσης του συναδέλφου Τίμωθη Κέρχο να αναμεθεί στην Ελλάδα. Και θα το συζητήσουμε σε μία από τις επόμενες Επίσης είπε πριν ο πρόεδρος ότι η έκθεση των πεπραγμένων στην αποστολή στην Ελλάδα αναβάλλεται. Επίσης έχουμε έναν κοινό τριμερή διάλογο όσον αφορά της κατεξοδότησης πράξης και σε σχέση με, το, με, όλα τα, με αυτές τις πράξεις που έχουν σχέση με το πολιετές πλαίσιο. Και αυτό θα συζητηθεί στις 26 Ιουνίου 4.30 με 6.30 το απόγευμα. Και θα ζητηθούν όλοι οι πόροι που έχουν σχέση και τα ταμεία που έχουν σχέση με την Επιτροπή μας. Ε, θα συμμετάσχουν οι συγκητές και σκιώδες και επίσης οι Επίτροποι Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Προχωρούμε τώρα, είναι το πρώτο σημείο ουσίας και έχουμε την ε, παρουσίαση. Α, όχι, όχι, όχι, λέει ο Πρόεδρος. I escaped. Ε, first... με. Αλλά πήγα παρακάτω, κατά λάθος, γιατί έχουμε τώρα το θέμα της προστασίας του ευρώ και άλλων νομισμάτων ε, δύναμη των διατάξεων του ποινικού δικαίου. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Άνθια Μακεντάιρ. Έχουμε επίση εδώ ε, μια, ένα σχέδιο οδηγίας. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά πάντοτε. Έγινε η παρουσίαση. Now we're going to hear the presentation of the draft report by Mrs. Μας παρουσιάζουμε στο σχέδιο της έκθεσης στο παρελθόν, κυρία McIntyre. Εκτός από το ενίο νόμισμα πάντως. Το θέμα είναι και η σημασία αυτού του μέτρου για την παραχάραξη παγκοσμίω. Κύριε Μακίντερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως προαναφέρατε, το θέμα είναι η προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων μέσω των διατάξεων του ποινικού δικαίου. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί, κωδικοποιεί τα ισχύοντα νομοθετήματα. Πρόκειται για σοβαρό έγκλημα εδώ, πρόκειται για παραχάραξη, για χαρτονομίσματα και ε, κέρματα. Και μιλούμε για ζημία ετησία 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι ετησίω από τότε που θεσπίστηκε το πρώτο 2002. Επομένω, θεωρούμε πάρα πολύ θετική αυτή την πρόταση. Δεν έχει επιμάχα σημεία. Έχουμε πάντω δύο σημεία στην έκθεση τα οποία παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα. Πρόκειται για τα σημεία που θα σα αναπτύξω δεν έχει τονιστεί όσο πρέπει το πόσο σημαντική πτυχή του θέματος είναι η εδαφικότητα και επίσης οι ελάχιστες ποινές που θεσπίζονται. Οπότε, όσοι επιτοπλίστων αυτό το σχέδιο κειμένου εύκολα μπορεί να συγκεντρώσει τη γενική συνένεση και λόγω αυτού του χρονοδιαγράμματος αυτό το οποίο κάναμε ήταν οι σκιοδησηγητές να ε, συναντηθούμε πριν την παρουσίαση του σχεδίου κειμένου. Και κάποια στιγμή υποπίεσε Είπαμε ότι ίσως μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τις τροπολογίες, εμείς οι σε εκείνη τη συνέντευξη, οπότε τελικά αφού τα συμφωνήσουμε όταν υπάρχει αδικημένο να μην κατεβάσουν τροπολογίες. Δεν αυτό δεν το καταφέραμε, αλλά πάντως ε, ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι μπορέσαμε οι σκιοδεσυγητές να τα συμφωνήσουν τα περισσότερα. Οπότε αυτό το σχέδιο εκθέσεως που τώρα έχουμε είναι σαν κείμενο πιο ουσιαστικό και από ό,τι φαίνεται πιο εύκολα θα συγκεντρώσει τη Γενική Συνένεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους σκιώδησηγητές και κυρίως τον κύριο Ντιόν για το έργο του, για την συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα, οπότε και έτσι. Οι πρώτες αντιδράσεις των εισηγητών ήταν το ότι θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι θα πρέπει να είμαστε αυστηροί με τέτοιου είδους ε, εγκλήματα. Και έλεγα λοιπόν ότι η αρχική αντίδραση ήταν αυτή, ότι πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι θα είμαστε πάρα πολύ αυστηρή με αυτό το έγκλημα. Όμως υπήρξε από τον κύριο Γιώργο και από μένα ε, η αμφιβολία το ότι δεν θα πρέπει να θεσπίσουμε ελάχιστες ποινές. Οπότε το σχέδιο έκθεσης που θα σας ε, πω έχει τις εξής βασικές τροπολογίες. Πρώτα πρώτα έχουμε την τροπολογία 1 και την τροπολογία 5 ε, έχουμε την τελική παράγραφο 23 και την παράγραφο 1 του άρθρου 8 σχετικά με αυτές τις τροπολογίες. Και θέλω να σας πω ότι βασικά θέλουμε να έχει αρμοδιότητα το κράτος μέλος εκεί όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Είναι καλύτερα. παρά να, τα κράτη να επιδιώκουν ε, την ε, τιμωρία αυτών που παρεχάρισαν νομισμά τους κάπου αλλού. Τώρα για τις ελάχιστες ποινές ε, θέλω να διαγραφεί μια ολοκληρή παράγραφος γιατί θεώρησα ότι αποτελεί επικάλυψη τροπολογίας. Όμως έχουμε το αρχικό κατόφλι των 10.000 ευρώ για ε, εγκλήματα, κολάσιμα με φυλάκιση 8 ετών. Και ε, επομένως είπαμε ότι έχουμε αυτό το κατόφλι των 5.000 ευρώ τώρα. Και μεγίστη ποινή φυλάκισης 8 έτη. Αλλά διαγράψαμε την ελάχιστη ποινή. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δικαστές εκείνοι να διαμορφώνουν την ε, κρίση τους. Γιατί η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οπότε με την ελάχιστη ποινή θα ήταν σαν να θεσπίζαμε διαφορές μεταξύ κρατών μελών, διαφορετική ποινική μεταχείριση. Και ελπίζω ο κύριος Ντεγιόν θα συμφωνήσει ότι τελικά είναι θέμα ε, του κάθε δικαστού, του κάθε κάθε ενόμης τάξης. Αυτές είναι βασικές αλλαγές. Επίσης, έχουμε και άλλη μια καινούργια τροπολογία, σύμφωνα με την οποία είπαμε ότι παραχάραξη ε, θα μπορεί να, με, με αφορμή παραχάραξη θα μπορεί να προσφύγει το κράτος μέλος στην συνεργασία με την όλα. Οπότε, με αυτές τις ε, παρατηρήσεις αυτές θα σας αναφέρω σε σχέση με την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κυρία Μακιντάρη. Να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Η κυρία Στρέφλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την ησυχήτρια για την εξαιρετική δουλειά της ε, και για την έκθεσή της. Όπως είπε, είναι το δεύτερο νόμισμα το ευρώ στον κόσμο και είναι στόχος των εγκληματικών ε, οργανώσεων παραχάραξης. Ε, αυτό βέβαια ε, σημαίνει τουλάχιστον 500 ε, εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες από το 2002. Ε, Η απειλή παραμένει πάρα πολύ σοβαρή, οπότε εγώ επικροτώ τη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να δημιουργήσει ένα κοινό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία Πρέπει να έχουμε μια συνεπή προσέγγιση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ποινικό δίκαιο. Πολλά κείμενα αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση στο Κοινοβούλιο, ειδικότερα η πρόταση οδηγίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν και το αντικείμενο μιας ε, συνεδρίασής μα της Θα είμαι σύντομη, γιατί όλα τα είπε η συγγήτρια σε σχέση με τις ελάχιστες ε, κυρώσεις. Εγώ πιστεύω ότι η επιβολή τους ε, ε, με τον τρόπο που, το, που αναφέρεται δεν είναι ο σωστός τρόπος γιατί ο δικαστής είναι αυτός που μπορεί κάθε φορά να σταθμίσει την σοβαρότητα του αδικήματος. Οπότε αυτά θα ήθελα να πω μόνο γιατί τα υπόλοιπα τα είπε η συγγήτρια. Ευχαριστώ και πάλι. Ο κύριος De Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της ως τώρα και για τη συνεδρίαση που είχαμε με τους σκιώδεις εισηγητές στο Στρασβούργο. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες από την ομάδα μου. Νομίζω ότι μπορώ να ακολουθήσουμε, μπορώ να ακολουθήσουμε την προσέγγιση σας. Ε, θα διαβάσουμε πολύ προσεκτικά το κείμενο, μπορεί να ζητήσουμε κάποιες αλλαγές διατύπωσης, αλλά η γενικότερη προσέγγιση της εισηγήτριας μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Ε, και το ΕΛΚ το είπε μόλις, υπάρχει μια σχέση βέβαια με την άλλη συζήτηση που κάναμε χθε σε σχέση με την οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και είδαμε ότι και σε αυτό το σημείο ε, εισάγει ελάχιστες κυρώσεις η Επιτροπή. Είχαμε τη συζήτηση εδώ χθε, ε, ήταν και αντιπρόεδρος ε, Ρέντινγκ μαζί μας. Το συζητήσαμε λοιπόν για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το βρίσκω λιγάκι ανησυχητικό ότι μία ακόμη φορά χρειάστηκε να εξηγήσουμε στην Επιτροπή ότι αν, αν ε, υπάρξει η έννοια των ε, ελάχιστων κυρώσεων, Είτε μα αρέσει είτε όχι, εμένα δεν μου αρέσει για πολλού λόγου, αλλά αν το αφήσουμε αυτό κατά μέρο, ακόμη και αν κάποιο είναι υπέρ, πρέπει να αναγνωρίσει ότι το σύστημα ε, ποινικού δικαίου είναι ένα σύστημα και αυτό που κάνει συστηματικά η Επιτροπή είναι να εισάγει νέε ιδέε συνεχώ σε μία, στη την άλλη πρόταση. Αυτό ακριβώ ε, ζητήσαμε ε, ω κοινοβούλιο στο παρελθόν να μην γίνεται. Οπότε περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα που έχει την αρμοδιότητα στον τομέα του ποινικού δικαίου να δείξει ότι είναι υπέρ μιας συνεκτικής και συνεπούς προσέγγισης για το ποινικό δίκαιο. Αν θέλετε να εισάγετε ε, ελάχιστες κυρώσεις, πρέπει να δείτε όλο το φάσμα των αδικημάτων και πού θέλετε να επιβάλλετε κοινώσεις, γυρώσεις. Ε, να πείτε ας πούμε ότι αυτό είναι το ε, ζήτημα του οικονομικού συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν αποτελεί από μόνο το επιχείρημα γιατί είναι σαν να δείχνει η Επιτροπή ότι δεν γνωρίζει πώς δουλεύει το έγκλημα ε, πώς δουλεύει το ποινικό δίκαιο. Μπορούμε να έχουμε μια καλή συζήτηση από αυτού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την προσέγγιση που έχει επιλέξει. Τελευταίο σημείο Κύριε Πρόεδρε, για τη συζήτηση που κάναμε χθε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για την λειτουργία τη Όλαφ, ε, η Όλαφ είναι πολύ σημαντική και για αυτή την έκθεση και νομίζω ότι θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες ε, που θα εκφράζουν ε, ανησυχίε σε σχέση με το πώς δουλεύει η φωτογραφία γραφείο καταπολέμησης της απάτης γιατί τα πράγματα έχουν αρκετά κλιμακωθεί. Για παράδειγμα εχθές με το ΕΛΚ και τους πράσινους να ζητούν την αποχώρηση του διευθυντή τη Όλαφ και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην μας διαφεύγει όταν ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Ο Πρόεδρο. ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μηπω θέλουν να σχολιάσουν. Η Ιόλαφ αν παρίσταται, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι από τη Γενική ε, Διεύθυνση Προϋπολογισμών. Θα ήθελα να πω ότι εγώ συμφωνώ ε, με αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε την παρακράτηση του ευρώ και άλλων ε, νομισμάτων πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, κάτι το οποίο με φέρνει σε αυτό που υπόθηκε για δύο ζητήματα. Πρώτον, το θέμα της καταλληλότητας του καθεστώτος ε, κυρώσεων για την παραχάραξη του ευρώ και το δεύτερο είναι ένα ζήτημα του ε, ποια δικαιοδοσία πρέπει να ισχύει. Για τις ελάχιστες κυρώσεις ε, γνωρίζουμε βεβαίως ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πρέπει να συζητηθεί ε, σε βάθος, όπως υπόθηκε άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπέρ μια συνεπούς και συνεκτικής ε, ε, πολιτικής για το θέμα αυτό, κατόπιν της ανακοίνωσής της του 2012. Κάτι ακόμη είναι σημαντικό, που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, όταν βλέπουμε για παράδειγμα τα αδικήματα, και την προσέγγιση μας επ' αυτού. Υπόθηκε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια συνεκτική γραμμή αν ακολουθεί μια συνεκτική γραμμή, γιατί για κάποια ε, θέματα όπως η προστασία των οικονομικών συμφερόντων υπάρχουν ελάχιστες κυρώσεις, ενώ για άλλα όχι. Εμείς αυτό δεν το βλέπουμε ως αντίφαση ε, που να πλήττει τη συνοχή της ευρύτερης πολιτικής, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να δούμε ε, τα καλά που προστατεύουμε με το ποινικό δίκαιο. Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά μεταξύ της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ε, και του ευρώ. Κατά τη γνώμη μας χρειάζεται, ε, πρέπει τα γνήσια ευρωπαϊκά προϊόντα να έχουν προστασία σε ολόκληρη την Ευρώπη και άλλες εγκληματικές πράξεις που είναι διασυνοριακού χαρακτήρα είναι επίσης σημαντικές βέβαια. Οπότε Αυτά σκεφτήκαμε και προ, προτείναμε ελάχιστες κυρώσεις για να ε, αντιμετωπίσουμε αυτά τα προϊόντα μεγάλης σημασίας που θέλουμε να προστατεύσουμε και δεν βλέπουμε ε, καμία διαφορά ή διάκριση όταν πρόκειται για σοβαρότερα δικήματα. Να πω μία ακόμη φορά ότι ελάχιστες κυρώσεις δεν είναι κάτι το αυτόματο. Υπάρχουν ανησυχίες ότι κάτι τέτοιο ε, θα σημαίνει ότι οι δικαστές θα είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν ελάχιστες κυρώσεις. Αυτό είναι κάτι βέβαια το οποίο απευθύνεται στο νομοθέτη αλλά όχι στα διάφορα δικαστήρια. Οπότε δεν βλέπουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ανησυχία. Και τέλος αυτό που είπε η κυρία Μάκενταρ για την ε, αρχή της ε, εδαφικότητας Υπάρχει ήδη ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και πολιτικές στο πλαίσιο αυτού και πιστεύω ότι πρέπει να βασιζόμαστε σε δύο κριτήρια, είτε το κριτήριο της εδαφικότητας ή ε, της εθνικότητας. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να μειώσουμε το πεδίο ε, εφαρμογής της δικαιοδοσίας των κρατών μέλων. Οπότε θα θέλαμε να σας ζητήσουμε επ' αυτού να διατηρήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη τις αρχές της εθνικότητας και της εδαφικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Το Συμβούλιο είναι εδώ. Θέλει να σχολιάσει. Όχι. Ο κύριος Μπρόγκ θέλει να πάρει το λόγο πριν θέσουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Όπως ε, ακούσαμε, είμαστε όλοι φυσικά κατά της παραχάραξης. Ακόμα και σε ό,τι αφορά το ευρώ, το τρισκατάρατο. Είχα την ε, εντύπωση ότι η παραχάραξη ήταν ε, έγκλημα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχει κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία να μην αποτελεί ποινικό αδίκημα η παραχάραξη. Αν η απάντηση είναι αρνητική, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο πρόβλημα υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται, θέλουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία, εναρμόνιση, ε, χωρίς κάποιο σκοπό, έτσι μόνο για το να υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή και επίσης να πούμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφαλώς δεν ε, επηρεάζει καθόλου ε, κράτη τα οποία δεν υπόκειται στο διεθνές δίκαιο. Σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες κυρώσεις τώρα, υπάρχουν κάποια στοιχεία στα διάφορα νομικά συστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με πολύ λίγες ε, εξαιρέξεις, ε, μάλλον πέρα από τα εγκλήματα τύπου φόνο, τύπου δολοφονία λόγω μέθης, ε, δεν υπάρχουν ελάχιστες ε, προδιαγραφές, ελάχιστα τέτοια πρότυπα. Οπότε δεν βλέπω γιατί να πρέπει να υπάρξουν εδώ. Η κυρία Μακιντάρ, λέει ο πρόεδρος, αν θέλει να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια, προσδιορίσουμε το, την προθεσμία για τις τροπολογίες. Ναι, εν συντομία. Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να την ε, καθησυχάσω είναι το εξής. Στην έκθεσή μου δεν έχουμε αφαιρέσει τη δυνατότητα δίωξης από κράτη-μέλη των ε, υπηκών του σε άλλες χώρες. Απλά αναφέρουμε τη θέση ότι η εθνική εδαφικότητα θα πρέπει να έχει να προέχει. Είναι πολύ μικρή η αλλαγή. Απλά δηλώνουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχεί ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του και όντε εισηγητέ για τη συνεργασία του, την οποία και εκτιμώ ιδιαίτερω. Ευχαριστώ. Νομίζω τώρα λοιπόν ότι μπορούμε να ορίσουμε την προθεσμία για τι τροπολογίε 10 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε για το σχέδιο έκθεση, το οποίο μόλι παρουσίασε η κυρία Μακεντάρη, η οποία είναι η συγγήτρια. Και τώρα λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το 4, την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης από τον Έλληνα Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Δέντια. Σε δύο λεπτά καταφτάνει ο Υπουργός. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα λοιπόν. Περιμένουμε τον Υπουργό. Παρακαλώ να μείνετε στην αίθουσα. As we said, no need for recess. We welcome most warmly. Καλωσορίζουμε. πολύ θερμά τον Έλληνα Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας των Πολιτών, τον κύριο Δενδιά, για να μας παρουσιάσει το, εθνικό σχέδιο, το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης για το άσυλο και τη μετανάστευση. Ξέρετε ότι έχουμε τακτικές επαφές με, είπα τους εκπροσώπους των κρατών μελών που ασχολούνται με το άσυλο, τη μετανάστευση, το, τα σύνορα, τον έλεγχο και τη διαχείρισή τους. Και προσπαθούμε να συντονίσουμε τις δραστηριότητές μας και τη διαχείριση των ταμείων. Ο Έλληνας Υπουργός είναι ευπρόσδεκτος για να μας παρουσιάσει το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης και στην συνεχεία θα δώσουμε το λόγο για συζήτηση. Μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε εδώ, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εκ των προτέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν είδη εισαγωγή, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε εσά και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μου δίνει την ευκαιρία να επεκταθώ σε ένα θέμα που για τη χώρα μου, την Ελλάδα και για την Ευρώπη, αν μου επιτρέπετε, είναι κομβική σημασία. Και αυτή η ευκαιρία για μας, για την ελληνική κυβέρνηση, για μένα και για το Υπουργείο μου είναι μεγάλη σημασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Η υποστήριξή σας, η κατανόησή σας και οι επικρίσεις σα ακόμα, αν μου επιτρέπετε, είναι τεράστια σημασία για μας. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μια ευσύνοπτη εκδοχή της ομιλίας μου, γιατί το πιο σημαντικό είναι οι δικές σας παρατηρήσεις και ερωτήσεις και όχι το να εκφράσω και να εκφωνήσω μακροσκελείς λόγους. Από τελευταία επίσκεψη που κάνετε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2012 έχουν γίνει πάρα πολλά. Πολλά επιτέθησαν για την πολιτική της Ελλάδας για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών στο Δουβλίνο παρουσιάσαμε τον αναθεωρημένο ελληνικό σχέδιο για τη διαχείριση ασύλου και μετανάστευσης που πιστεύουμε ότι είναι μια ανθρώπινη αποτελεσματική απάντηση της κυβέρνησής μας στις σημερινές προκλήσεις του ασύλου και της μετανάστευσης. Στο φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης και στα θέματα που επηρεάζουν τους λαθρομετανάστες. Περί τίνος πρόκειται. Τι δημιουργήθηκε από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι σήμερα, που ήταν η τελευταία σας επίσκεψη στην Ελλάδα και που είδατε επί τόπου πώς έχουν τα πράγματα. Πρώτον, τα κέντρα υποδοχής. Η πρώτη υπηρεσία υποδοχής, η υπηρεσία πρώτης υποδοχής, ε, ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάρτιο του 2015 και θα γίνει πλήρως λειτουργική, λειτουργεί ήδη, αλλά μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα είναι απόλυτα λειτουργική. Επίσης, δύο ακόμα τέτοια κέντρα πρώτης υποδοχής ε, φτιάχνονται στη Λέσβο, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Αττική, το νομό που είναι πρωτεύουσα η το νομό της πρωτεύουσας και θα είναι ε, πλήρως λειτουργικά μέχρι το τέλος του 2013. Ε, συνεργαζόμαστε με την ε, ύπατη αρμοστία Ελλάδος, με ψυχολόγους, με... υπάρχει μετάφραση, διερμηνία. Επίσης, έχουμε δύο κέντρα προελέγχου, στη Χίο και στη Σάμο, που έχουν επανα... επαναδροθεί και είναι λειτουργικά από φέτος. Επίσης έχουμε... έχουμε... Είμαστε στη διαδικασία επάνδρωσης δύο κινητών μονάδων. Γιατί? Γιατί ο τρόπος και τα μοντέλα της λαθομετανάστευσης αλλάζουν. Πριν είχαμε το πρόβλημα του Εύρου, τώρα έχουμε το πρόβλημα του Αιγαίου. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να προσαρμοζόμαστε. Δημιουργούμε λοιπόν αυτές τις δύο κινητές μονάδες. Επίσης, για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο φαινόμενο, εγώ ανέλαβα από το Υπουργείο Εργασίας και Δημόσιας Υγείας την υπηρεσία που προσφέρουμε προς τις ευπαθείς ομάδες. Και δημιουργήσαμε δύο κέντρα για αυτές τις ευπαθείς ομάδες στην Αθήνα, και σχεδιάζουμε δύο ακόμα. Επιλέξαμε τα μέρη που θα τα στεγάσουν και θα είναι ε, λειτουργικά και αυτά μέχρι το τέλος του 2013. Στις αίρες το ένα, ε, Κεντρική Μακεδονία. Και ένα ακόμα. Το άσυλο στην Ελλάδα ήταν ένα αντικείμενο τεράστιων συζητήσεων και η νέα αρχή ασύλου της Ελλάδας έχει δημιουργηθεί, λειτουργεί στα νέα της γραφεία στην Αθήνα και η νέα αρχή προσφυγών επίσης υπάρχει και λειτουργεί στα νέα της γραφεία στην Αθήνα. Πέραν αυτών, θέλουμε τα πέντε κέντρα τα περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Οριστιάδας και Ρόμπου να τα επανδρώσουμε. Ε, για τον Εύρο και για, το πρόβλημα του Εύρου και την, ε, το Αιγαίο και θα είναι επιχειρησιακά σύντομο. Α, υπάρχει ένα κέντρο από τις 7 Ιουνίου λειτουργικό που έχει, έχει λάβει 63 ε, αιτήσει από γυναίκες, 9 από ανήλικους ε, και 144 από άντρες. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε επίσης και τις καθυστερημένες υποθέσεις τις παλιές υποθέσεις. Όταν ανέλαβα το περασμένο Ιούλιο, είχαμε 55.000 που δεν είχαμε διεκπαιρέωση για το άσυλο. Τι κάναμε με αυτές τις υποθέσεις. Δημιουργήσαμε καταρχάς ένα ηλεκτρονικό κέντρο, ψηφιοποίησαμε όλους τους φακέλους και τις, τους 55.000 φακέλους. Και από την ηλεκτρονική μορφή αρχίσαμε τη διεκπαιρέωση. 17.000 ε, ε, διεκπαιρεώθηκαν και από τις υπόλοιπες. Ε, οι 3.606 είχαν ήδη εκδικαστεί και για να διπλασιάσουμε την ταχύτητα ε, διπλασιάσαμε τις επιτροπές που ασχολούνταν με τις καθυστερημένες υποθέσεις. Από 10 φτάσαν σε 20 σε στενή συνεργασία με την ε, υπατιαρμοστία προσφύγων Ελλάδος. Τα προαναχωρησιακά κέντρα. Δημιουργήσαμε πέντε κέντρα προαναχωρησιακά, Μυγδαλέζα τον Οκτώβριο ήδη όταν επισκεφθήκατε το είχαμε ε, με 200 θέσεις. Τώρα έχουμε πάνω από 1.500 θέσεις στην Κόρδο, Κομωτινή, which is... το Παρανέστη, ε, ένα στην Αττική, ένα στην Πελοπόννησο και τα τρία τελευταία είναι στη Βόρεια Ελλάδα η συνολική χωρητικότητα ξεπερνάει τις 5.000 θέσεις. Το σχέδιό μας είναι να δημιουργήσουμε 10.000 θέσεις. Και έχουμε επιλέξει παλιά κέντρα τα οποία μπορούν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν και να γίνουν προαναχωρησιακά κέντρα. Έχουμε τις κλασικές τα κλασικά πρότυπα με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση την ελληνική εθνική νομοθεσία λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών για τον καθαρισμό, την ασφάλεια, τον ανεφοδιασμό σε τρόφιμα, ε, υπάρχει διαγωνισμοί οι οποίοι ε, δρομολογούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το ποιος θα αναλάβει αυτά τα έργα. Η ανάγκη δημιουργίας αυτών των κέντρων οφείλεται στο ότι υπάρχει πρόβλημα και κόλλημα στις επιστροφές. Ο θέμα στο οποίο θα επιστρέψουμε μόλις ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση που εξελίσσεται με την Κομισιόν για το ποιος μπορεί να πάει σε ένα τέτοιο προαναχωρησιακό κέντρο. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε να σας πω ότι κατά τη γνώμη μας ότι με το να αναζητήσουμε τι κάνει το άσυλο, να επιδιώκει το άσυλο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει ελεύθερος και κυκλοφορών στην Ελλάδα. Πολλοί λαθρομετανάστες καταχρώνται το δικαίωμα ασύλου υπό την εξή έννοια. Δεν υποβάλλουν το αίτημα ε, ασύλου κατά την είσοδό του στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επομένω. Υποβάλλουν αυτή την αίτηση μόλις, μόνο όταν συλληφθούν από την αστυνομία σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ε, μια απλή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι αυτοί οι άνθρωποι που τότε υποβάλλουν την αίτησή τους ε, καταχρώνται του συστήματος. Έχουμε μια τεράστια συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι πρακτικό. Φαίνεται ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ μακριά. Δημιουργούμε λοιπόν ένα μηχανισμό με βάση τον οποίο όλοι, όλες οι υποθέσεις ασύλου που αφορούν άτομα που είναι ήδη σε κράτηση θα εκδικαστούν μέχρι τον Αύγουστο του 2013, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες από σήμερα. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν σε μια ενδιαφέρουσα νομική συζήτηση. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία για την... Καμία ουσία μάλλον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Οι επιστροφές. Ένα τεράστιο θέμα. Ξέρετε ότι κάποια εγκαταστάσεις έχουν ε, κλείσει, έχουμε κλείσει την Βένα, το ελληνικό, τον ασπρόπυργο, το τυχερό και έχουμε αλλάξει την ε, εγκατάσταση του ελληνικού η οποία όμως θα κλείσει και η καινούργια εγκατάσταση που μάλλον μέσα στο 2013. Οι επιστροφές τεράστιο θέμα, πολύ σημαντικό. Υποστηρίζουμε υποστηρίζουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα που δρομολογήθηκε τον Αύγουστο του 12 για τον εθελοντικό επαναπατρισμό για να ε, στείλουμε πίσω άτομα τα οποία εκδόσαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν από μόνα τους και μέσω του, της διεύθυνσης επαναπατρισμού η ελληνική αστυνομία ε, εφαρμόζει ένα δικό της πρόγραμμα επιστροφών. Όμως, όπως και να έχει το πράγμα, οι επιστροφές, οι επαναπροωθήσεις είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί, για έναν απλό λόγο, γιατί, γιατί οι βασικές χώρες προέλευσης δεν συνεργάζονται μαζί μας. Αναφέρομαι ειδικά στο Αφγανιστάν, στο Μαγκλατές, στο Πακιστάν, στο Ιράκ, στην Αλγερία και στο Μαρόκο. Αυτές οι χώρες είναι περίπου το 80% του προβλήματος. Ζητήσαμε τη βοήθεια της Κομισιόν για να πιέσει αυτές τις χώρες και πέρα από τις συμφωνίες επανεισδοχής, πέρα από την υπογραφή τους ή στην περίπτωση που υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες επανεισδοχής, να τις εφαρμόσει. Και οφείλω να σου ομολογήσω ότι δεν είναι ικανοποιημένο με την κατάσταση. Και ούτε με την πίεση που ασκείται σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι επαρκής. Έλεγχο των το τελευταίο κεφάλαιο. Είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στην περιοχή του Εύρου, που ήταν το μείζον πρόβλημά μας. Έχουμε δύο επιχειρήσεις, ένα εξέλιξη, Ξένιος Δίας και την επιχείρηση Ασπίδα. Να σας δώσω ένα νούμερο. Μία μέρα πριν από την έναρξη της επιχείρησης Ασπίδα, 412 λάθρομετανάστες διέλευσαν τον Εύρο. Και τώρα περίπου τρεις ή τέσσερις τη βδομάδα λαθομετανάστες περνάνε τον Εύρο. Φυσικά έχουμε πρόβλημα στο Αιγαίο. Το Αιγαίο δεν αποτελεί ευθύνη δική μου, του Υπουργείου μου, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι και εδώ δημιουργούμε ένα σύστημα με βάση το οποίο τα ευρωπαϊκά σύνορα του Αιγαίου θα προστατεύονται. Με μια επιχείρηση που θα την ονομάσουμε μάλλον Ποσειδώνα. Αλλά ένας άλλος υπουργό θα έρθει να σας ενημερώσει για τα σχέδιά μας για το Αιγαίο. Είναι κατακλείδη. Σας προσκαλώ ακόμα μια φορά να επισκεφτείτε την Ελλάδα το φθινόπωρο που μας έρχεται μετά την περσινή σας επίσκεψη και να δείτε η διεισόμαση, την πρόοδο που πετύχαμε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δένδια, για την ε, παρουσίαση του ελληνικού προγράμματος δράσης όσον αφορά την διαχείριση των μεταναστευτικών ορών. Τώρα έχουμε ε, τα μέλη της Επιτροπής που θα αναλάβουν το λόγο. Οπότε ε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια το ότι έχουμε και ψηφοφορία, μην το ξεχνάτε αυτό, διότι ως συνήθως πρόκειται να έχουμε πάρα πολύ δουλειά, θα, θα, έχουμε όλο αυτό το, το, το στρες του να τρέχει ο κόσμος μέσα έξω με τις, ε, ε με τις κάρτες για να ψηφίσει. Ένα δίλεπτο παρακαλώ ο καθένας, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και, τα... και, και παρατηρήσεις προς τον κύριο Υπουργό. κυρία Ματιώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό που ήρθε να μας παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα δράση όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Έτσι μπορούμε να ενημερωθούμε όσον αφορά τα προβλήματα αυτά τα οποία αναδύονται μέσω των αιτήσεων ασύλου, γιατί έχουμε αυτά τα προβλήματα με την μετανάστες και το άσυλο. Ακούσαμε πάλι προσεκτικά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, της Πρόεδρος, που σημείωσε η κυβέρνησή σας όσον αφορά την, την πρώτη υποδοχή τους ε, συνοδεύτους ε, ανηλίκους και επίσης έτσι μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ε, τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των ετούντων άσυλο και βλέπουμε ότι όλα αυτά σιγά σιγά εξομαλύνονται και βεβαίως μπορούμε να αισθανθούμε κάποια ικανοποίηση. Επίσης μας είπατε τι γίνεται με αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό Ακόμη βέβαια έχουμε κάποια σημεία που παρουσιάζουν πρόβλημα, ε, τα προβλήματα για την χρηματοδότηση. Οπότε και βεβαίως εμείς μπορούμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε ε, να βοηθήσει τη χώρα σας. Επίσης θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς η κατάσταση θα εξομανηθεί γενικότερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πιέσει και το Συμβούλιο όσον αφορά τον επανεντοπισμό των ε, ετούντων του άσυλου. Να δούμε πώς θα υπάρχει κάποιο είδου κατανομή του, της δουλειάς του έργου που πρέπει να επιτελεστεί. Θα πρέπει κάτι να γίνει, θα είπαμε και ότι η χώρα σας έχει αναλάβει όλο αυτό το βάρος και υπάρχει βεβαίως μία δυσφορία ακριβώ γιατί ε, είναι δεδομένος ο πληθυσμός της χώρας και δεδομένο επίσης το πόσο είναι αυτοί που ζητούν άσυλο. Οπότε θα πρέπει να πιαστεί το Συμβούλιο για να βοηθήσει. Και να δούμε κατά πόσο να ξανασυνθεί το ζήτημα στην Ολομέλεια, κύριε Υπουργέ. Ο πρόεδρο. Και τώρα για να δούμε η ελληνική αντιπροσωπεία. Α, πρώτα πρώτα ο κύριος Μούλτερ. Η αντιπροσωπεία μας στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι από τότε που επισκεφθήκαμε την Ελλάδα, ακούγοντα τον ε, κύριο Υπουργό, έχουμε σημαντικέ βελτιώσει. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε παρά να το θεωρήσουμε πάρα πολύ θετικό. Το είχα πει τότε και δημοσία ότι με εντυπωσιάζει η νοοτροπία, η στάση των ε, υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν ε, αυτό το πρόβλημα με τόσο δύσκολες συνθήκες υπό την συγκυρία της κρίσης. Οπότε, γι' αυτό και το σούτο μάλλον θεωρούμε ότι είναι επένετη αυτή η βελτίωση. Γι' αυτό και το είπαμε και δημοσία. Τώρα, έχουμε κάποια σημεία που ακόμα μας ε, προβληματίζουν. Έχουμε αυτά τα κέντρα κράτησης. Εκεί οι συνθήκες επιδέχονται βελτίωση, δεν είναι και Είχαμε πει ότι ε, μέχρι την 1η Απριλίου θα πρέπει να έχουν κλείσει κάποια αυτά τα κέντρα κράτησης. Δεν κατάλαβαν αυτό ε, έγινε ή όχι. Θα ήθελα να με ενημερώσετε κύριε Υπουργέ. Και Αν σας καταλάβω καλά κύριε Υπουργέ, ε, και με τους ετούντες στο άσυλο και εκεί έχετε βελτιώσει την κατάσταση. Βέβαια το πρόβλημα αυτό σώβει και στην Ελλάδα και αλλού στην Ευρώπη και έχουμε επίσης πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε καθεστώς γκρίζο το πούμε. Είναι παράνομοι και δεν είναι και παράνομοι. Είπαμε θα περάσετε σε ψηφιοποίηση, ό,τι σημαίνει αυτό. Διαπέστε πέστε μας ακριβώς τι θα κάνετε όσον αφορά ε, αυτούς όλους τους ανθρώπους. Θέλω κι άλλο να ρωτήσω, αλλά θα βάλω εδώ τελεία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Πίρκερ, μία παρατήρηση καταρχάς. Ε, ήμασταν στα σύνορα υπό την καθοδήγηση του κυρίου Μούλτερ με την ομάδα μας και είδαμε όλοι μαζί πώς είχε η κατάσταση, παρακολουθήσαμε τα πράγματα, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα πράγματα. Ακόμα πιο ενδιαφέρον ήταν ότι είχαμε μία έκθεση για τις ε, παρατηρήσεις μας. Η έκθεση αυτή ολοκληρώθηκε πριν από κάποιες ημέρες και απευθύναμε στον πρόεδρο της Επιτροπής. Δεν ε, είδα σε καμία επιτροπή τέτοιες εκθέσεις ε, μίας επίσκεψης, μίας, ε, μίας ε, αποστολής να κάνουν τόσο χρόνο να ολοκληρωθούν. Μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή βλέπουμε ότι παραλείπονται λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται τόσο πολύ χρόνος για να ολοκληρωθούν τέτοιες εκθέσεις. Δηλαδή, οι βουλευτέ οι οποίοι έχουν κάνει μια αποστολή να χρειάζεται να περιμένουν ολόκληρου μήνε για να δουν την έκθεση αυτή, μου φαίνεται πραγματικά πολύ περίεργο. Αυτό λοιπόν, Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσω, θα σας παρακαλούσα να φροντίσετε, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Τώρα στις, σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις σας. Η Ελλάδα αναμφίβολα αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και στο παρελθόν αλλά και σήμερα ακόμα. Και σε καμία περίπτωση δεν ήταν προετοιμασμένοι για όλες αυτές τις εισρωές οι οποίες ήταν αναμενόμενες και οι οποίες εμφανίστηκαν. Όπως και ο κ. Μιόλτερ, πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ θετική η εντύπωσή μου σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ρωτώ, λοιπόν, ποιες είναι οι επιπτώσεις των επενδύσεων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των συνόρων. Είδαμε σε ό,τι αφορά την έγερση του φράχτη, ε, συνεργασία με τη Frontex, όλα αυτά είχαν επιπτώσεις. Καταπολέμησαν την ε, εγκληματικότητα αυτή, καταπολέμησαν το γεγονός ότι άλλαξαν για παράδειγμα οι διαδρομές ε, εισόδου λαθρομεταναστών. Και κάτι άλλο, μια δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά τους έτοντες άσυλο. Μιλήσαμε με πολλούς ετούντες άσυλο, μάλλον με πολλά άτομα τα οποία ήταν σε αυτά τα κέντρα και σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να κάνουν αίτηση για άσυλο, αλλά ότι ήταν εκεί για οικονομικούς λόγους. Έχει αλλάξει αυτό. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ε, αιτήσεων για άσυλο. Σημαντικά. Μιλήσατε επίσης για το ότι πολλοί κάνουν αίτηση για άσυλο μόλις συλληφθούν από την αστυνομία. Έχετε κάποια στοιχεία για το χρονικό διάστημα για το οποίο παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι ότου να συλληφθούν και μέχρι ότου να κάνουν την αίτηση για άσυλο. Ύστερα, στις διαδικασίες για άσυλο όταν τελικά απορριφθεί μια τέτοια αίτηση για άσυλο, ποιες είναι οι συνέπειες. Λειτουργούν οι επιστροφές. Τους δέχεται η χώρα προέλευσης, όπως αναφέρεται και προηγουμένως. Πρέπει μέχρι τις 10.30 να ψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ να το έχετε υπόψη, να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε σε δύο λεπτά. Εντάξει, θα δείξουμε φυσικά κάποια επίοικια, αλλά σας παρακαλώ να θέσετε τις ερωτήσεις σας. κύριε κύριο Πονικολάου. Θα μιλήσω πολύ. Και εγώ από την Ελλάδα είμαι, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω λοιπόν σήμερα. Κάποιες ερωτήσεις κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε. Αναφερθήκατε το θέμα, στο θέμα της χρηματοδότησης. Πώς έχει σήμερα ακριβώς η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την Ελλάδα. Η Επίτροπος Μάλμστρομ στην Επιτροπή αυτή, ξέρετε, έρχεται συχνά και συνηθίζει να λέει ότι εξακολουθεί να υπάρχει χρηματοδότηση. Εγώ, εξ όσων γνωρίζω, έχουμε προβλήματα χρηματοδότησης στην Ελλάδα. Πώς έχει λοιπόν η κατάσταση ακριβώς και τι προσδοκά και η ελληνική πλευρά. Τι περιμένει η ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Μαράμ Η κυρία Γκυγιώμ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ πιο σύντομα για να μην καθυστερούμε να κερδίσουμε χρόνο. Εγώ συμμετείχα στην ε, ε, επίσκεψη στην Ελλάδα. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Πίρκερ σε σχέση με την ταχύτητα της ε, έκθεσης αυτής, διότι υπάρχουν πολλές πιέσεις, αντιφατικές για να το πω έτσι, από πλευράς όλων. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με την ε, βία για την οποία έχουμε ακούσει ότι υπάρχει στην Ελλάδα ε, σε σχέση με κάποιους μετανάστες ε, σε κάποια σημεία της Ελλάδας και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για τους μετανάστες εργαζόμενους, ποια είναι η άποψή σας για τη βία εναντίον των ανθρώπων αυτών και πώς μπορούν να επιληθούν αυτά τα προβλήματα βίας, με ποιον τρόπο. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την ενημέρωση που μας ε, έχετε παράσχει. Εγώ ήθελα να σας πω το εξής. Λόγω του αριθμού των προσφύγων, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες φέτος στη χώρα σας, μας είπατε ότι μιλούμε για 144 και 63 γυναίκες εξ αυτών. Με αυτά τα κέντρα κράτησης, τι γίνεται. Το πρόβλημά σας είναι αυτοί οι 55.000 υπαλλοί. Τι θα, πώς θα τους διαχειριστείτε είπατε. Ε, τα είπαμε στην Επιτροπή. Και έχουμε 17.000 ε, ε, οι οποίοι έπρεπε να υποστούν κάποια, κάποια μεταχείριση και το 2012 μας λέει η Eurostat ότι μόνο η Γαλλία είχε 96.000 αιτήσει. 37.000 στο Βέλγιο, ε, η Σουηδία 47.000. Μόνο το 2012, μιλούμε τώρα για τα στοιχεία της ε, Eurostat. Οπότε, το πρόβλημα είναι εσείς τι προποδότηση έχετε, τι προϋπολογισμό έχετε για όλους αυτούς. Ε, γιατί μιλούμε για τρίμηνα, για εξάμηνα και αυτοί απελευθερώνονται και μετά όμως ξαναγυρίζουν στα κέντρα κράτησης. Επομένως, τι θα γίνει με την ε, χρηματοδότηση, με την πρικοδότηση, γιατί συνεχίζουν τα προβλήματα με την ε, Τουρκία και έχετε λοιπόν όλε αυτές τις αρχές που ασχολούνται με την υποδοχή αυτών όλων των προσφύγων. Επομένως υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης και με αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται στα κέντρα κράτησης. Και ε, σα το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι στο Νότο υπάρχει αυτό το πρόβλημα παντού και στη δική μου χώρα την Ισπανία. Οπότε. Να, ποια είναι η διαφορά με τι χώρε του, του Βορρά. Ζητούμε ελληνική, αλλά εμεί στι χώρε του Νότου δεν αναγνωρίζουμε τόσο πολλού από αυτού που ζητούν το άσυλο του αναγνωρίζουμε ω πρόσφυγες. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Θα μπορούσαμε να του στείλουμε αλλού, αυτού όλου, θα μπορούσαν να πάνε αλλού, αλλιώς κάθονται στις χώρες μας μέχρι ότου ε, νομιμοποιηθούν. Βλέπω όλα αυτά τα στοιχεία της Eurostat και βλέπω ότι συνεχίζει να σοβεί αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν μπορείτε να το επιλύσετε. Θα λυθεί με την ευρωπαϊκή βοήθεια. Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Μήπω θα πρέπει να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια επίλυση. Δεν ξέρω. Έχετε του εμπειρογνώμονε που χρειάζονται τόσο ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε αυτού που έρχονται. Ε, Μπα και πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με την Τουρκία. Γιατί από Αλγερία, από Μαρόκο, όλοι αυτοί που πάνε να μπουν στην Τουρκία δεν του αφήνουν η Τουρκία. Δεν του δίνουν ε, θεώρηση διαβατηρίου. Επομένω, μία φορά να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του εδώ, όπως επίσης και για τη θερμή του υποδοχή όταν τον Οκτώβριο επισκεφθήκαμε την Ελλάδα. Βέβαια το είχαμε κάνει και παλαιότερα. Τον Οκτώβριο είδαμε ότι υπήρξε πολύ καλή πρόοδος και από ό,τι άκουσα σήμερα ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος έχει σημειωθεί και σας συγχαίρουμε γι' αυτό θα ήθελα να πιστεύω ότι οι περιορισμοί που είχατε για την πρόσληψη προσωπικού λόγω της Τρόικας έχουν αρθεί σε σχέση με τις υπηρεσίες, ώστε η νέα υπηρεσία ασύλου να μπορεί να είναι ε, σωστά επανδρομένη και ε, λειτουργική. Θα ήθελα τώρα να περάσω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και είναι το θέμα ε, της επανεγκατάστασης ε, των δικαιούχων ε, διεθνούς προστασίας. Έχουμε συγκεκριμένες διαδικασίες και αν τηρούμε σωστά τις διαδικασίες, όταν αναγνωρίζεται ένας πρόσφυγας ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, δεν μπορούμε να τους πανεντάξουμε στις κοινωνίες μας. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι ε, ένα σύστημα επανεγκατάστασης και ρωτήσαμε σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας είπε ότι τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν επ' αυτού. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο στο Συμβούλιο έχετε καμία πρωτοβουλία για να πείσετε τα κράτη-μέλη να δεχθούν την πρότασή μας ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει η ειδική πρόταση για ένα σύστημα επανεγκατάστασης το οποίο θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να μοιράζεται τις ευθύνες. Ευχαριστώ. Κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. Θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης η οποία δέχεται την μεγαλύτερη μεταναστευτική η πιο μεγάλη πίεση μέσα σε όλη την Ένωση. Επίσης, έχει τα πιο εκτεταμένα σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα. Μιλώ και κατά και βέβαια και από πλευράς θαλάσσης και ακτών. Πρόκειται επομένως πραγματικά για το εξωτερικό σύνορο της Ένωσης. Και επισημένω την πολύ σημαντική οικονομική προσπάθεια που καταβάλει η Ελλάδα με αυτό το πρόγραμμα δράσης. Επισημένω ότι πρόκειται βέβαια για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε αυτή την τόσο περίπλοκη οικονομική συγκυρία. Οπότε και θέλω να καταλήξω στο ότι θα πρέπει να επισημάνουμε τα δύνατα σημεία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Και τελικά μία λέξη μου έρχεται στο μυαλό αλληλεγγύη, αλληλεγγύη ευρωπαϊκή προς την Ελλάδα. Αυτή η αλληλεγγύη βεβαίω θα πρέπει να συνοδεύεται από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την ε, επιστροφή και τον, την επαναπρόθεση. Και όσον αφορά τα κέντρα κράτησης. Ουσιαστικά όλα τα κεντρικά της τα επισκεφθήκαμε σε εκείνη την αποστολή. Και επομένως με την αλληλεγγύη θα πρέπει να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί φυσικά παντού υπάρχουν προβλήματα. Το Αιγαίο είναι η πιο σημαντική πύλη εισόδου στην ε, Ευρώπη. Από εκεί έχουμε τις πιο σοβαρές ε, ροές λάθρομετανάστευσης. Έχουμε επομένω αυτέ τι επιχειρήσει που τώρα λαμβάνουν χώρα, τις δύο σημαντικέ επιχειρήσει που λαμβάνουν χώρα και κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό το οποίο ε, είναι σημαντικό είναι να ξέρουμε τι κάνει η Frontex. Δεν είναι θέμα στρατηγική ανάλυση, δεν είναι θέμα συγκρηματοδότηση όσον αφορά τι νόμιμε επαναπροωθήσει δεν αρκεί να έχουμε κοινέ επιχειρήσει όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Αυτό το οποίο θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη είναι ότι εμεί σαν Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσουμε και θα πρέπει επίση και η Ελλάδα μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που, που βρίσκεται τώρα και από πλευρά μεταναστευτική θα πρέπει να αναγνωριστεί το ότι καταβάλει τεράστιε προσπάθειες και ότι θα πρέπει να τη βοηθήσουμε γιατί από μόνα τη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Μα, ξέρουμε ότι και η Μάλτα έχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά φυσικά διαφέρει πάρα πολύ η περίπτωση τη Μάλτα και από πλευρά έκταση τη νήσου και από πλευρά πληθυσμού. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κύριε Δρότσα. Ευχαριστώ πολύ. να μιλήσω στα ελληνικά. Κύριε Υπουργέ, να σα καλωσορίσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα και να σας συγχαρώ για ένα τόσο ελπιδοφόρο σχέδιο δράση για το άσυλο και τη διαχείριση τη μετανάστευση και σίγουρα αν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε κατά γράμμα αυτό το σχέδιο θα αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας. Δυστυχώς γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας στην Ελλάδα δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι η εφαρμογή του εκάστοτε σχεδίου και όχι η εκπόνησή του και να είστε σίγουρος ότι όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές θα κάνουν ό,τι μπορούν για να έχετε την αναγκαία στήριξη από την Ευρώπη για να εφαρμόσετε αυτό το σχέδιο. Θα σας ζητήσω όμως, αν μου επιτρέπετε, να μας βοηθήσετε και εμάς προχωρώντας τάχιστα στις απαραίτητες αλλαγές, στερώντας έτσι επιχειρήματα εναντίον της ε, Ελλάδας. Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό και ο φίλος Ισπανός ε, συνάδελφος μόλις ε, το τόνισε, το βάρος για την Ελλάδα είναι δυσανάλογο. Το γνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα, ελπίζω να το γνωρίζουν και οι εταίροι μας. Δεν μπορεί να τιμωρείται μια χώρα επειδή αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ε, Ένωσης ή βρίσκεται κοντά σε εστίες ε, κρίσης. Για μας είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει η αλληλεγγύη, η αλληλεγγύη πρέπει να είναι αυτονόητη. Η οικονομική βοήθεια βεβαίως είναι σημαντική και σε κάθε παρέμβασή μας δεν ξεχνούμε και να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την οικονομική βοήθεια που δίδεται στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από την Επιτροπή, αλλά δεν μπορεί η οικονομική βοήθεια να είναι το μόνο. Πρέπει να υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη. Για μένα αυτό είναι ηθικό θέμα, είναι και θέμα των αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω αυτό να αναγνωριστεί ακόμα περισσότερο από τους εταίρους μας και να είστε σίγουρος ότι σε κάθε παρέμβασή μας και στην Ολομέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς αυτό το τονίζουμε. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε και κύριε Πρόεδρε, ζητώ την κατανόησή σας λίγα δευτερόλεπτα ακόμα να τελειώσω την παρέμβασή μου με την εξής παρατήρηση ότι η διαχείριση της μετανάστευσης περνάει από μια επιτυχημένη πολιτική ενσωμάτωση των μεταναστών σε μια χώρα και ένας βασικός, ίσως ο βασικότερος πυλώνας μιας επιτυχημένης ενσωμάτωσης είναι να υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων και τελικά ηθαγένεια, ώστε οι μετανάστες που ζουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα να είναι ενσωματωμένοι στην πολιτική μας κοινότητα. Ξέρω ότι το θέμα της ηθαγένειας δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά οι συνέπειες της έλλειψης της σας ε, αγγίζουν άμεσα, γι' αυτό αναρωτιέμαι κύριε Υπουργέ γιατί η σημερινή κυβέρνηση πολέμησε τον νόμο περί θαγένειας που για πρώτη φορά έδινε κάποιες λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Δέκα και μισή έχουμε τη δυσκολό, το δυσκολότερο κατάλογο ψηφοφορίας και υπάρχουν ακόμη συνάδελφοι που θέλουν να, ε, να θέσουν ερωτήματα και πρέπει να έχει χρόνο και ο Υπουργός να απαντήσει. Δύο λεπτά έκαστος. Ε, yes. Κυρία Ινετφέλτ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ε, καλωσορίσω θερμότατα τον Υπουργό. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι έχουμε τη δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδας, όχι λόγω της οικονομικής κατάστασης, αλλά λόγω και, και της γεωγραφικής της θέσης. Ε, θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απογοητεύσει την Ελλάδα σε σχέση με την αλληλεγγύη που θα ε, έπρεπε να δείξει σε πολλού τομεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η Ελλάδα δεν έχει τι ευθύνε τη ε, όσο αφορά την σωστή πολιτική ασύλου και μετανάστευση. Δύο ερωτήματα λέτε ότι υποστηρίζετε το, το την αρχή της συστηματικής κράτησης ετούντων άσυλο. είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον ένα, ένα ε, κόμμα της Ολλανδικής κυβέρνησης ε, φαίνεται να το υποστηρίζει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα απορρίψουμε. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι πρέπει να κρατούνται άνθρωποι που δεν είναι εγκληματίες. Δεύτερον, ε, η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει οι επιστροφές ε, ετούντων άσυλο στο ελληνοτουρκικό σύνορο. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Ε, δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε αν ε, το θέμα αφορά μόνο το άσυλο και τη μετανάστευση. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για τη δημόσια τάξη. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Μιλάμε για άσυλο και μετανάστευση λέει ο Πρόεδρος. Αν έχετε λίγο χρόνο να μου απαντήσετε πάντως θα ήθελα να μου πει ο υπουργό τι κάνει σε σχέση με τη βία ε, της Χρυσής Αυγής. Thank you very much. Η κυρία Κέλλερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ, που ήρθατε εδώ και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει κάποια πρόοδος. Είναι πολύ κοινικό, ωστόσο, αυτό που λέτε για την κατάχρηση του συστήματος ε, ασύλου. Γιατί λέτε ότι υπάρχει κατάχρηση, αλλά για ποιο άσυλο μιλάμε. Είπατε κι εσείς ότι ε, είναι σχετικά πρόσφατη αυτή η υπηρεσία για αίτηση ασύλου και δεν είναι λοιπόν περίεργο το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση τώρα γιατί και εμείς ως πράσινοι πήγαμε στα κέντρα κράτηση στην Αθήνα και δεν υπήρχε τρόπο ο, ο κόσμος να ζητήσει άσυλο. Άρα πώ λέτε να ζητάει ο κόσμο κατευθείαν άσυλο όταν δεν μπορεί να το κάνει γιατί πρόκειται για ένα δικαίωμα ξέρετε δεν είναι έγκλημα αυτό και αυτή η ιδέα κράτηση ε, των ετούντων άσυλο ή έστω να υπάρχει και μια τέτοια δυνατότητα. Θεωρώ ότι καταπατά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Κάποιες ερωτήσεις. Πώς ε, εξετάζετε λοιπόν τα θέματα και πώς ε, διαμορφώνεται και το προσωπικό σε ό,τι αφορά τις αιτήσει άσυλο και πόσο παίρνει μια αίτηση για άσυλο και πόσο χρόνο παίρνει μέχρι να πάρει κανείς μια πρώτη απάντηση στην αίτηση αυτή. Είπατε ότι έχετε 17.000 φακέλους και αιτήσει για άσυλο και τις έχετε επεξεργαστεί ήδη και ότι θα κάνετε και πιο πολλά μέχρι τον Αύγουστο. Πώς θα το κάνετε αυτό διασφαλίζοντας παράλληλα και τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Και για πείτε μας, και δεν γίνεται με το ποσοστό αναγνώρισης, γιατί η απόφαση του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έλεγε ότι ε, θα πρέπει να ισχύουν και οι σχετικές προδιαγραφές για την αναγνώριση των προσφύγων στην Ελλάδα και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το ποσοστό αναγνώρισης. Και τέλος, σας είχαμε γράψει ήδη το Νοέμβριο ως πράσινη μία επιστολή αναφορικά με την κατάσταση στην Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τα κέντρα κράτησης. Ακόμα δεν έχετε απαντήσει. Δύο λεπτά ο για κολλήνω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος. Χαιρόμαστε για την πρόοδο για την οποία μας μίλησε ο Υπουργός. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η παρουσίασή του. Μας μίλησε για τους συνόδευτους ανηλίκους, για, για τους χρόνους διεκπαιρέωσης. Την περασμένη εβδομάδα ε, ε, υιοθετήσαμε και τον κανονισμό του Δουβλίνου και το πακέτο για το άσυλο. Εμείς ως ε, Ιταλική αντιπροσωπεία δεν ήμασταν σύμφωνοι, όπως δεν ήταν και η ελληνική αντιπροσωπεία, γιατί δεν υπάρχει αλληλεγγύη, γιατί δεν επιμεριζόμαστε σωστά το άχθος. Επίσης, θα πρέπει όλα τα κρατη να συμμετέχουν και όχι μόνο εκείνα τα οποία υφίστανται τρομακτική μεταναστευτική πίεση όπως η Ελλάδα σε αυτό το σύστημα. Επίσης, το επιστησιακό σχέδιο της ε, Frontex είχε σαν σκοπό να υποστηρίξει συγκεκριμένα τα άτομα τα οποία ε, στη χώρα προέλευσής τους ε, διώκονταν, κινδύνευε η ζωή τους και χρειάζονταν λοιπόν προστασία. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τις τεράστιες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Στην Ελλάδα βέβαια υπάρχει το πρόβλημα του Αιγαίου. Σε πολλά άλλα κράτη που έχουν και αυτά μεταναστευτικές ροές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της Μεσογείου εν γέννη. Επομένως θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό προστασίας που θα ήταν πολύ χρήσιμος για το θέμα της Μεσογείου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε ευχαριστώ. Η πολιτική σημερινή απλή αποδοχή ότι οι χώρε έχουν δυσκολίε και έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τα ταξιδικά του έγγραφα έχει να κάνει με το χαμηλό ποσοστό επιστροφών και αυτή η προσέγγιση που είναι λανθασμένη αποστέλει ένα μήνυμα το οποίο θα ήταν προς τους λαθρομετανάστες ότι είτε θα τους αφήσουν να μείνουν είτε θα τους αρνηθούν το δικαίωμα αλλά και πάλι θα μπορούν να μείνουν περιμένοντας τα, τα έγγραφα τα οποία ποτέ δεν φτάνουν μετά από χρόνια, μετά από μήνες ε, και δικαστικές αποφάσεις ή αλλιώς θα περιμένουν ε, να εισακουστούν οι αιτήσει του. Αυτοί οι παράγοντε προσελκύουν όλο και πιο πολλού λαθρομετανάστε που προσπαθούν να δοκιμάσουν την τύχη του και οι χώρε προέλευση καθυστερούν ή και αρνούνται να εκπληρώσουν τι ε, ευθύνε του σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή των επικών του. Αυτέ λοιπόν θα πρέπει να κατανομαστούν και θα πρέπει να του ασκηθεί πίεση να αποδεχτούν τι ευθύνε του και αν ε, συνεχίσουν να αποτυγχάνουν η Ελλάδα και άλλε χώρε θα πρέπει να δώσουν μονομερείς άμεσες ε, βοήθεια, αν θέλετε, στις ε, ε, ανθρώπους αυτούς να επιστραφούν στις χώρες τους. Γιατί η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο μέσα σε ένα τεράστιο πρόβλημα με τους περιορισμούς που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Αλλά φυσικά είναι και αυτή τμήμα του προβλήματος. Η επιχείρηση Ασπίδα, όπως μας είπαν, έχει μεριορίσει τις εισρωίες, ε, τις μεταναστευτικές, κατά 6,9%. Η εντύπωση που δίδεται είναι ότι η χώρα προσπαθεί να επιλύσει ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά αντιμετωπίζει μια τεράστια πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί της επιβάλλει υποχρεώσεις ε, και έτσι η οικονομία μπορεί να πλήττεται από τη λιτότητα η οποία επιβάλλεται από μια διάφορη Ευρωπαϊκή Ένωση και η ταυτότητά της υποσκάπτεται από το μεταναστευτικό θέμα, από τις μεταναστευτικές εισρωές. Ευχαριστώ. Μίσης Κύριε Υπουργέ, ε, αντιλαμβάνομαι και ανησυχώ όπως και πολλοί συνάδελφοι για το γεγονός ότι με την εφαρμογή του Δουβλίνου 2 θα δημιουργηθούν τρομακτικά προβλήματα στις πύλες εισόδου των μεταναστών. Την άλλη ανησυχώ και για τα ενδεχόμενα προβλήματα τα οποία θα υποστούν οι ήδη οι διακινούμενοι και αναρωτιέμαι αν ένα από τα μέτρα για, τον ισότιμο, για την ισότιμη κατανομή του βάρους δεν θα ήταν με την εφαρμογή και του readmission agreement η επιστροφή αυτού που θα αποστέλνεται στην Ελλάδα, στη Μάλτα, στην Κύπρο ενδεχομένως κατευθείαν στην χώρα από την οποία έχει εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθούσε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Chrysogoulos. Κύριος Χρυσόγελος. Yes. Yes, please. Ε, κύριε Υπουργέ, ε, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σίγουρα χρειάζεται η Ευρώπη να δείξει μεγαλύτερη ελεγγύη και να μην υποκρίνεται, αλλά και η χώρα μας δεν έχει κάνει πολλά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Πριν από λίγες μέρες επισκεφθήκαμε μαζί με τη συμπρόεδρο της ομάδας των Πράσινων, την κυρία Ρεμπέκα Χάρμ, στο κέντρο κράτηση που υπάρχει στην Αμυγδαλέζα. Βέβαια, η χώρα μας θα, θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει κέντρα υποδοχής και όχι κέντρα κράτησης. Αλλά σας αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που εντοπίσαμε στα κέντρα κράτησης Υπάρχει άτομο, ενδεικτικά είδαμε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει άτομο το οποίο έχει πιστοποίηση βασανιστήριων. Είναι στο κέντρο κράτησης για πάνω από 7-8 μήνες και ξέρετε ότι κάποιος που έχει βιώσει βασανιστήρια, όταν κρατείται, ε, ξαναζεί αυτή την εμπειρία. Υπάρχει πιστοποιημένο από άτομο το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Προέρχεται από το πρώην κέντρο αποκατάστημάτων βασανιστήριων. Δεύτερο άτομο είναι, έχει αδελφή που έχει άδεια παραμονής και δικαιώματα στην Ισπανία. Δεν έχει επανενωθεί με την αδελφή του και είναι πάνω από 7-8 μήνες μέσα στο κέντρο κράτησης. Ε, υπάρχουν άτομα τα οποία προέρχονται από το Ιράν και έχουν κάνει αίτηση για άσυλο. Είναι μέσα πολλούς μήνες ό,τι προέρχονται από το Ιράν και δεν έχουν ε, ακόμα απαντηθεί τα ερωτήματά τους προς το άσυλο. Επίσης, δίπλα από το κέντρο κράτησης ενηλίκων υπάρχει κέντρο κράτησης ανηλίκων. Πολλές περιπτώσεις, αλλά σας αναφέρω μία ενδεικτική. Νέος που κατάγεται την Αλβανία, 17,5 χρονών, ήρθε στην Ελλάδα ενός χρόνου, τα υπόλοιπα 16,5 χρόνια ζει στην Ελλάδα, μιλάει μόνο ελληνικά, πηγαίνει στο σχολείο και κρατείται σε αυτό το κέντρο και θα πάρει σε 6 μήνες ελληνική ταυτότητα. Και τέλος είναι το θέμα της θαγένειας. Πολλά άτομα είναι μέσα 16 και 17 χρόνια στα κέντρα κράτη, 16 ε, και 17 χρόνια στην Ελλάδα, παρόλα αυτά είναι στα κέντρα κράτησης αυτή τη στιγμή. Καλώ Παπαδόπουλου. Παπαδοπούλου. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Η ερώτησή μου αφορά ακριβώ ε, την κοινοτική αλληλεγγύη. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι τρομακτική η μεταναστευτική πίεση στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Νότο, όπω και στη, Μεσέ, με, στη, στη Μεσόγειο και διερωτούμε πραγματικά αν υπάρχει σωστός καταμερισμός βαρών ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε αυτό το κοινοβούλιο διαρκώς λέμε ότι αυτές τις πιέσεις από αιτητές ασύλου, λαθρομετανάστες και μετανάστες, τις δέχεται κυρίως ο Ευρωπαϊκός Νότος που αντιμετωπίζει παράλληλα την οικονομική κρίση. Και μια δεύτερη ερώτηση όσον αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου λάθρο μεταναστών και δυστυχώς διοχετεύονται από τα σύνορα εις τον Εύρο. Ε, τι στήριξη θέλει η Ελλάδα ώστε τα δημοκρατικά λύματα που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά ε, και τα υπηρεσιακά σχέδια της Frontex αλλά και στη συνεργασία των χωρών αυτών να βελτιωθούν. Πώς μπορεί να στηρίξει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελευταία, ε, θα πρέπει να πω ότι υποστηρίζω και εγώ τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προστασία, ειδικά για τι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου και τη Μεσόγειο, γιατί είναι διαφορετική η πίεση που δέχονται αυτέ οι χώρε συγκριτικά με άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you, colleagues. Please, Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ λίγη ησυχία, γιατί ε, ο Υπουργό πρέπει να έχει χρόνο να απαντήσει σε όλα αυτά τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Υπάρχει το θέμα της αλληλεγγύης. Ε, ενδιαφέρον βέβαια έδειξαν πολλά μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Να προσθέσω και εγώ την ε, δική μου προσωπική συμπόνια ε, συμπάσχω πραγματικά με το ιδιαίτερα εκτεθειμένο εξωτερικό σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, που είναι υπό την αρμοδιότητα της Ελλάδας. Παρακαλώ να σας πω, να σας θυμίσω, ψηφίζουμε στις 10.30. Σας ζητώ λιγάκι υπομονή, γιατί πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός στα ερωτήματα που του ετέθησαν. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη, μου προς την Επιτροπή σας που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω εδώ και για το ενδιαφέρον σας, για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την Ελλάδα. Το, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να απαντήσω ερώτηση προς ερώτηση, αλλά δεν μου επιτρέπει ο χρόνος που έχω. Επομένως, ας κάνω μια συνοπτική, ας δώσω μια συνοπτική απάντηση σε όλα τα θέματα. Τον περασμένο Ιανουάριο υποσχεθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο δράσης. Αυτό το σχέδιο δράσης το από ένα κέντρο υποδοχής, πρώτο κέντρο υποδοχής, το οποίο είναι λειτουργικό με ένα νέο σύστημα ασύλου, το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή, με ένα νέο, νέα αρχή προσφυγών, υπάρχει και αυτή, και μία πολιτική επαναπροώθησης ή επιστροφών η οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, με ρωτήσατε και τα παλιά ε, προαναχωρησιακά κέντρα. Ο κύριος Μούλντε με ρώτησε που ήταν στην Αθήνα με μέλη της Επιτροπής σας να σας απαντήσω ότι αυτά τα κέντρα που επισκεφτήκατε εσείς εκτός από ένα δεν υπάρχουν πια. Το ελληνικό έκλεισε, το παλιό ελληνικό έκλεισε και το νέο ελληνικό, αυτό που επισκεφθήκατε εσείς, δεν υπάρχει όπως το είδατε. Ε, έχει αλλάξει και θα κλείσει το άλλως με αυτό το 2013. Για τις παλιές ε, υποθέσεις ε, ασύλου που δεν έχουν διεκπαιρεωθεί, που με ρωτήσατε, Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να... Αυτοί που έχουν διεκπαιρεωθεί ε, δεν θέλουν να ξανανοίξουν οι ενδιαφερόμενοι και από τις υπόλοιπες 3.606 ε, το ποσοστό διεθνούς προστασίας που έχει δοθεί είναι 25,28%. Για το θέμα της Τουρκίας, η Τουρκία προσπαθεί να αλλάξει, αλλά δεν ε, λαμβάνουμε και την υποστήριξη που περιμέναμε. Ε, το 2012 υποβάλαμε στην Τουρκία σχεδόν 25.000 ε, αιτήσει επανεισδοχής και μόνο 113. 113 από αυτές, από όλα αυτά τα άτομα τα δέχτηκε η Τουρκία πίσω. Φυσικά υπάρχει το θέμα των οικονομικών δυσκολιών. Να σας δώσω τα νούμερα. Θα δώσω και μια, ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή, ούτω ώστε όλοι να δείτε τα νούμερα. Αλλά το συνολικό κόστος του νέου σχεδίου ανά έτος είναι περίπου 5 δις. Από αυτά 250, 247 για την ακρίβεια, τα δίνει ο ελληνικός προπολογισμό. Η ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι 178 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε ευγνώμονε, αλλά είναι λιγότερο από αυτό που δίνει ο ελληνικός προϋπολογισμός για την ε, λαθρομετανάστευση. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, μεγαλύτερη στην ελληνική ιστορία. Και ε, μας λείπουν 72 εκατομμύρια. Μιλήσαμε με την Επιτροπή. Η Κομισιόν προτείνει να χρησιμοποιήσουμε ε, τα ποσά που έχουμε στη διαθέσή μας. Τα έχουμε απορροφήσει όλα και τώρα μας προτείνει η Κομισιόν να χρησιμοποιήσουμε τα διαφορετικά ταμεία. Τα διαφορετικά ταμεία δίδονται σε προτιμησιακή βάση. Επομένως δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εύκολα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κάνουμε, ιδίω για να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Προσπαθούμε, αλλά φαντάζομαι ότι φοβάμαι ότι η χρηματοδότηση είναι επαρκή. Μιλάμε για ένα ύψο, συνολικό πόσο 500 εκατομμυρίων ε, ευρώ. Και ένα τεράστιο θέμα για μας επανεγκατάσταση. Οτιδήποτε και να κάνουμε κύριε και κύριοι πρέπει να συζητηθεί μεταξύ μου Ευρωπαίων. Ό,τι και να κάνουμε κάποιοι όμως πρέπει να επαναγκατασταθούν. Εμείς είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορούμε να απορροφήσουμε 500-600 χιλιάδες λαθρομετανάστες. Δεν μπορούμε. Απλούστατα όπως η Γερμανία δεν μπορεί να απορροφήσει 10 εκατομμύρια φερρυπίν λαθρομετανάστες. Χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Πρέπει να εγγύψει στο πρόβλημα. Πρέπει να δει το πρόβλημα. Και θα πρέπει να αρχίσει τη συζήτηση για ένα, θέμα, για ένα θέμα που θα έπρεπε να είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και εμεί, λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μα διαθέσατε, για τις προσπάθειές σας για να δημιουργήσετε αυτή τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης που μας παρουσιάσατε. Σας ευχαριστούμε. And as we said... Και όπως είπαμε λοιπόν, Έχουμε και την ψηφοφορία τώρα. Σας παρακαλώ να προετοιμαστείτε λοιπόν για την ψηφοφορία. Σας υποστηρίζω το εξή. Ε, καταρχάς χρειαζόμαστε την κάρτα ψηφοφορίας. Έχετε όλες τις κάρτες σας. La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 Get Προετοιμαστείτε παρακαλώ, ξεκινάει η ψηφοφορία. Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, σα παρακαλώ, ξεκινάει η ψηφοφορία. Καθίστε, τι κάρτε σα να έχετε έτοιμε. Έχετε κανένα διαδικαστικό, κυρία Μόρβαϊ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ε, κάνω μια ερώτηση για την ημερήσια διάταξη. Χτες στις 11.30 λάβαμε ένα τμήμα της, ε, του καταλόγου ψηφοφορίας που χρειαζόταν μεγάλη επεξεργασία. Σήμερα στις 9.30 λάβαμε και, άλλες, ε, και άλλα έγγραφα, τα οποία και αυτά χρειάζονταν κάποια επεξεργασία. Και σήμερα το πρωί χρειάστηκε να πάμε και σε άλλη ψηφοφορία. Η έκθεση βάρες για την Ουγγαρία και την δημοκρατία για την Ουγγαρία αναφέρει σε μία παράγραφο ότι χρειαζόμαστε και χρόνο για την νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν ε, αγαπητοί βουλευτές θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς συνάδουν αυτά τα σημεία για το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Τι θέλετε να κάνετε προκειμένου να μην παρουσιαστούν τέτοια φαινόμενα πάλι στο μέλλον. Και κατά δεύτερον η έκθεση Ταβάρες, η έκθεση που συζητούμε σήμερα Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα αντίσταται στις δικτατορίες. Και πολλοί συνάδελφοι έρχονται εδώ και... Ε, σηκώνουν τέτοια συνθήματα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να υψώσω και την Ουγγρική σημαία θα ήθελα να επιμείνω και να πω ότι και εγώ έχω δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν είναι σημαντικά τα θέματα αυτά. Εσείς είσαστε αναφέρετε φασιστές ε, συνάδελφοι. Δεν νομίζω ότι σας επιτρέπω να με ονομάσετε φασιστρία. Να πάνε όλα καλά στην ψηφοφορία. Σας παρακαλώ ηρεμήστε, ησυχάστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε στις ε, ψηφοφορία. Όχι, όχι, δεν σα επιτρέπω να αναφέρετε τέτοια φασιστικά. Ναι, σα παρακαλώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο. Δεν, είσαστε, δεν είμαστε σε τσίρκο. Κάνουμε ψηφοφορία τώρα, λέει ο πρόεδρο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα πώ έχει η κατάσταση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι περίπλοκη η ψηφοφορία. Σα παρακαλώ, συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε παρακαλώ στην διαδικασία αυτή. Να έχουμε όλοι υπόψη ότι ε, μας πιέζει ο χρόνος, ότι έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες ε, εξέπρασης εμβιβασμών μεταξύ του εισηγητή και των σκιωδών. Είναι πολλές οι πολιτικές ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο. Κύριε Ταβάρες, δεν ξέρω αν θα θέλατε να μιλήσετε για ένα λεπτό πριν από την ψηφοφορία. Αν όχι, αν δεν θέλετε το λόγο, να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Θέλετε να πάρετε το λόγο, να κάνετε σχόλια για τις ε, προσπάθειες που έγιναν για εξέπρεση συμβιβασμού. Ναι, εν συντομία, να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες, όλους τους βουλευτέ που απέστειλαν τροπολογίε, που ε, εργάστηκαν σκληρά την έκθεση αυτή να σας μιλήσω και για τρεις πρόσφατες εξελίξεις που δεν αποτυπώνονται ακόμα πλήρως στην έκθεση αυτή. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την επίσημη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας που δημοσιεύτηκε μόλις πριν από δύο ημέρες για την Ουγγρική κυβέρνηση, για την απόσυρση της τέταρτης τροπολογίας στο Σύνταγμα και μία δήλωση της κυρίας Αναδίπηλα της είπα της αρμοστή για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λίγο πολύ τα ίδια είπε όπω και η Επιτροπή της Βενετία και όπως ξέρετε στην τελευταία συζήτηση για την Ουγγαρία ζήτησα από την Ουγγρική κυβέρνηση να μας δώσει επίσημη μετάφραση του νέου νόμου για την εθνική ασφάλεια το οποίο μας απασχολούσε γιατί θα έδινε την ευθότητα σε παρακολούθηση και υποκλοπή επαφών ε, δικαστών και εισαγγελέων και αυτό φυσικά καταπατά την διαχωρισμό των εξουσιών. Δεν μας έχουν ακόμη δώσει τη μετάφραση του σχετικού νομοσχεδίου. Θα δούμε κατά πόσον θα κάνουμε δική μας μετάφραση και όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην έκθεση και θα είναι έτοιμη η έκθεση για την Ολομέλεια. Να ευχαριστήσω όλους τους Ούγγρους πολίτες που μας έχουν γράψει. Τους απάντησα και κάποιοι έχουν απαντήσει και αυτοί με τη σειρά τους και έτσι έχουμε ξεκινήσει έναν πολύ καρποφόρο διάλογο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών που μας απασχολούν όλους. Και θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει ο και τώρα να επικεντρωθούμε στην ψηφοφορία. Γιατί θα πάρει χρόνο. Θα πάρει χρόνο. What is that? I mean, of course, of course, of course, of course, this, this, this cannot happen. This situation here. Έχετε δίκιο, δεν μπορεί να επιτραπεί αυτή η κατάσταση σας παρακαλώ στο τεχνικό ε, προσωπικό να ε, συμμορφωθεί. Δεν είναι τσίρκο εδώ πέρα, κυρία Μορβάη, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έπρεπε να ξέρετε κάπω καλύτερα τι επιτρέπετε και τι όχι πριν έρθετε στις, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα παρακαλώ λοιπόν να παρακαλήσω την τεχνική υπηρεσία να επικεντρωθούμε στην ψηφοφορία, να σταματήσουμε το τσίρκο αυτό, γιατί θα πάρει χρόνο η ψηφοφορία. Έχουμε πολλέ σελίδε ε, καταλόγου ψηφοφορία και κάποιες παράγραφοι θα πρέπει να ψηφιστούν μεμονωμένα παρά τις προσπάθειες εξέφρασης συμβιβασμού. Ναι, κύριε Βίξτρο, έχετε το λόγο. Πρόεδρε. Πρόκειται για εργασίες της Επιτροπής. Θα περάσουμε σε ψηφοφορίες και κάποιοι εξημών ημών έχουμε ενοχληθεί ιδιαίτερα από τις ανοησίες αυτές που επιδεικνύονται στην αίθουσα. Μας ενοχλούν ιδιαίτερως. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Να γίνεται ψηφοφορία με ζωντανή μετάδοση στο ίντερνετ, να το βλέπουν αυτά οι πολίτες στο διαδικτύο. Είναι απαράδεκτο. Ναι, ναι, φυσικά λέει ο Πρόεδρος. Χαίρομαι που καθαρίζουμε την αίθουσα και που αφαιρούμε τα περαιτά για την ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ασφαλώς λέει ο Πρόεδρος, το είπαμε αυτό ξεκάθαρα, ας είμαστε αξιοπρεπείς, παρακαλώ, και αποδίδοντας τον δέοντα σεβασμό στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ας συνεχίσουμε. Συμβαστική. Θα ανακοινώσω μία προσθήκη τελευταία στιγμή. Η τροπολογία 250 καταπίπτει εάν περάσει ο συμβιβασμός 9. Οι 2.66 και 2.67 επίσης καταπίπτουν αν εγκριθεί ο 24. Η 395 δεν καταπίπτει αν περάσει η συμβαστική 18 και η 154 καταπίπτει αν ο συμβιβαστική 41 περάσει. Μετά λοιπόν από τις ανακοινώσεις αυτές, η κυρία Ενσφέλτ θέλετε να πάρετε το λόγο. Εντάξει, ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για την ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, υπέρ. Η τροπολογία 195. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η παράγραφος 3. Τροπολογία 197. 98, 199. Α, συγγνώμη, 197 και 198. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την παράγραφο 3. The vote is open. Ένταξη ψηφοφορίας. Παράγραφ 3. Για την παράγραφο 3 λέει ο πρόεδρος. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Τι πρόβλημα υπάρχει. 190, 196, 197 197 και 198 στην παράγραφο 3. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Μα περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Τι πρόβλημα υπάρχει. Η 197 αφορά την παράγραφο 2 και όχι την παράγραφο 3. Όχι, ψηφίσαμε την παράγραφο 2 ήδη. Και ήταν η τροπολογία 195, τώρα ψηφίζουμε την 197-198 παράγραφος 3. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, μισό λεπτό. We're voting now. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την παράγραφο 2, την 195, πριν περάσουμε στην παράγραφο 3. Λοιπόν, να ψηφίσουμε την παράγραφο 2, την 195. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην παράγραφο 3. 100... Ναι, έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Έχω την εντύπωση ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ αν δεν αναφέρετε τις παραγράφους. Μόνο τους αριθμούς των τροπολογιών. Νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. And let's go only for the number of the amendments. Εντάξει, θα λέω μόνο τον αριθμό των τροπολογιών. Άρα, 197 και 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 201 και 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 206. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός στις 206. Τέρας της ψηφοφορίας. Είστε υπεράριθμοι στο ΕΛΚ. Δύο παραπάνω. Μείον δύο στο ΕΛΚ. Τι γίνεται. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ψηφισάντων του ΕΛΚ. Μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Για να δούμε τώρα. 39 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Από τη 208 στη 211. Τις ψηφίζουμε όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 214 και 15 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 222 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 236 έως 230... Α, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. 235, 236, 237 και 238, όλε μαζί τι ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. 239. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 240. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. Άρα πάμε στη συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 250 καταπίπτει. Πάμε στη 251 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική... Α, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται. Έκανα λάθος. Ήταν περισσότερα τα χέρια που είδα για κατά από ότι για υπέρ. Συγγνώμη, απορρίπτεται δικό μου το λάθος, λέει ο πρόεδρος. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει. Λοιπόν. Πέρα στις ψηφοφορίες. απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257, 258, 259, όλες μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 263 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 264, καταπίπτει, καταπίπτει. Ναι, αλλά η 262 έχει αποσυρθεί. Μα έχει αποσυρθεί η 262. Έτσι γράφει ο κατάλογος μου. Δικό σας τι λέει. Α, εντάξει. Λοιπόν, ψηφίζουμε Ψηφίσαμε τη 263 και απορρίφθηκε. Τώρα, αν θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 263. Ωραία, έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 263. Πέρα τη ψηφοφορία. 24 Απορρίπτεται. 264 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 272 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 277 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 278 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 280 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστη... Ε, συγγνώμη, 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 288 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 289 υπέρ κατά. Μ, δεν είναι σαφές. Δεν σηκώνετε καλά τα χεράκια. Ψηφίζουμε τη 289 ηλεκτρονικός έλεγχος ένερχη της, ένεξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη 289. Το ΕΛΚ υπεράριθμο κατά έναν. Πέρας της ψηφοφορίας. Σαφέστατα απορρίπτεται. Δεν σηκώσατε αρκετά τα χεράκια σας. Τέλος πάντων μπερδεύτηκα εγώ με τα χέρια. 292. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Α, να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τι. Τη 294. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 294 έναρξη ψηφοφορίας, πέρας της ψηφοφοριας 2331. 23-31. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. 310 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 311 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 313 Α, συγγνώμη, ήταν μαζί αυτές οι δύο τροπολογίες. 314 ε, υπέρ. 314, 315 πάνε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Πάμε στην 316. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Θέλετε να ψηφίσουμε τη 316 ηλεκτρονικά. Ωραία. Έναρξη ψηφοφορία για την 316. Πέρας. 23-31. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 317. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, έλεγχος. Ηλεκτρονικός της 317. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. «23-33 απορρίπτεται. Προχωρούμε. 318, όπως είπα προηγουμένως, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 320. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 321 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 321 καταπίπτει. Α, θέλετε να την ελέγξουμε την 321. Ωραία, να την ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Απορρίπτεται, απορρίπτεται σαφέστατα. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 325 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 327 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 329 υπέρ. Κατά. Έλεγχος, έλεγχος. Την 329. Γιατί υπήρξε σοβαρή αποχή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικό στην 329. Έναρξη ψηφοφορίας. Είναι 26-16. Με 16 εποχές. Εγκρίνεται. 330. Όχι. Α, όχι. 335 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 338 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 339 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 340 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 341 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 342 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 343 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 345 Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρι... Συμβιβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24. Υπέρ. Α. Αποχές. Εγκρίνεται. 366 τώρα. Α, καταπίπτει. Α, συγγνώμη. Λάθος τροπολογία. 368 τώρα. Το δεύτερο τμήμα που εξακολουθεί να ισχύει υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 375 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 376 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 377 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική 25 ηλεκτρονικός, να την ελέγξουμε. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. 33 ε, υπέρ, 23 κατά. Πάμε στην 395. Ε, Η προηγούμενη υιοθετήθηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Και προχωρούμε. Πού είναι? 449. 449. Πάμε στο 449. Απ, πήγαμε μερικε προσελίδε παρακάτω. 449. 449. Είναι δική μου αυτή η τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Ναι. Κύριε Έγγελ, καταλαβαίνω ότι θέλετε αυτό που θέλετε. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 449. Ψηφίζουμε. Πέρας. Τριάντα δεν Εγκρίνεται. Οριακό το αποτέλεσμα, αλλά εγκρίθηκε. 488. Δεύτερο τμήμα. 488. Το δεύτερο τμήμα. Τη βρήκατε. Σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην 500. Όχι, λέει ο Πρόεδρος. Έλεγχος στο δεύτερο τμήμα του 488. Πέρας. In. Και προχωρούμε τώρα. Abstentions rejected. Ε, απορρίπτονται. Συμβιβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 503. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική όχι, συγγνώμη, το πρόεδρος 504 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 505 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θα έχουμε κάποια προβληματάκια σε λίγο. Πάμε στο 522. 522. Όχι, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 519. 519. Βρήκατε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στο 521. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 521. Ψηφίζουμε. Πέρας. Είκοσι, απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στο 522 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 523 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος για το 522 καταμέτρηση πέρας 42-12 απορρίπτονται. 5.23 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Το ηλεκτρονικό έλεγχος για το 523. Ψηφίζουμε. εγκρίνεται. 5.25 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτα. 527. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτα. Συμβαστική 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την συμβαστική 29. Ψηφίζουμε. ο της 35-22 εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 42. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την συμβαστική 30. Ψηφίζουμε. 43-21. 42. Συμβαστική 42. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική 42. Ψηφίζουμε. Πέρας. Πέρας. 30-27. Οριακό, αλλά εγκρίνεται. Πέντε σαντένια. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέντε πενήντα. Υπέρ. Κατά. 5.50. Ελεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρας. 27.30. Απορρίπτωται. 5.51. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Όχι, δεν κατέπεσε. Άρα ορθός. και ψηφίσαμε. Ιδεολογικές παραγράφη τώρα. Αιτιολογίες παραγράφη. Ναι, μα ψηφίσαμε. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Ψηφίσαμε την 501. Την 551 μάλλον. Τώρα πάμε στις αναφορές και τις αιτιολογικές σκέψεις. Πρέπει να ε, ψηφίσουμε καταρχήν την τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές, ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε την τροπολογία 13. Γιατί δεν σηκώσατε τα χέρια. Ψηφίζουμε. της ψηφοφορίας. 39 υπέρ 17 κατά. Υιοθετείτε σαφώς. Πάμε στη 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 και 17 μαζί. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε 15. Αρχίζουμε τώρα. Πέρας της ψηφοφορία. 36 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Συγγνώμη κυρία Βεωζιά. Οι 16 και 17 ψηφίζονται μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Now compromise 31. Συμβασμός 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 19 και 20. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 και 22 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Εποχές υιοθετείται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 27. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 33 υπέρ Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. Συμβασμός 32. Περ. Κατά. εποχές, Υιοθετείται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Υπέρ. κατά, εποχές υιοθετείτε, 42 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείτε, 45 υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείτε, 46 υπέρ, κατά,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 Μπερδεύτηκα. Πάμε στο συμβασμό 35. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Διοθετείτε. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Πηδήξαμε μια τροπολογία του Έγγελς. Την 62. Ψηφίζουμε την 62. Υπέρ. Καταπίπτει. Λάθος, λάθος, μπερδεύτηκα. Κακός μου τα είπανε, κύριε Έγγελς. Κύριε Έγγελ. Την 63 ψηφίσουμε, όχι την 62. Την οποία ψηφίσαμε ήδη. Όμως. Να τζεκάρουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Και θετείτε. Πάμε στο συμβασμό 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 76. Υπέρ κατά, αποχές υιοθετείται, 38 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται, 81 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβασμός 82, 82, τροπολογία των διορθών των πρόεδρων. Τροπολογία 82 και όχι συμβασμός 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 88. Κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 καταπίπτει αυτό ε. όχι δεν καταπίπτει είναι ζωντανό το ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 40. Υπέρ. Κατά αποχές Υιοθετείτε. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 101. Favor. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 102. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά rejected. απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές διαθετείται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 114 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 117 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές διαθετείται 126 υπέρ κατά αποχές διαθετείται όχι απορρίπτεται συγγνώμη 127 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται, 128 υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείται, 129 υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείται, 130 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται, 131 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 132 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε, 133 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 134 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 135 και 36 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 137 και 138 ψηφίσμα μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 140 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 141 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 142 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 143 υπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ. 145 κατά. Αποχές 146 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 149 ηλεκτρονικός έλεγχος για να μην κάνουμε λάθη. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 26 κατά, 31. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 151, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ. 176. Δεν το έχω στον κατάλογο ψηφοφορίας μου. 176. Υπέρ. Δεν το έχω στο κατάλογο ψηφοφορίας μου, λέει ο πρόεδρος. Πρόβλημα, πρόβλημα. Δεν έχουν και οι σοσιαλδημοκράτες το 176 στον κατάλογο ψηφοφορίας τους. κατά λάθο έχει παραλευθεί από τον κατάλογο ψηφοφορίας με ενημερώνων. Όπως και να έχει, είναι της Κίνγκα Γκάλ και του Λάσλο Σούριαν. Η τροπολογία 176 θέλετε να σας διαβάσω. Να σας διαβάσω, λέει ο Πρόεδρος. No, listen, listen, listen. Ακούστε λοιπόν. Σκοπός ε, της τροπολογίας 176 είναι η διαγραφή της παραγράφου της εξής. Opinion, blah, blah, blah, of March 19 of the right on freedom of conscience and religion and the legal status of churches, denomination religious communities of Hungary. So, is a... Διαγραφή της παραγράφου λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτή την παραπομπή που γίνεται στην ε, Επιτροπή της Βενετίας. Ε, εντάξει, θέλετε να το ψηφίσουμε. Ωραία, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν τώρα στην 177. Το ίδιο. Η ίδια κατάσταση. Τροπολογία Φρανκ Έγγελ. Διαγραφή και πάλι. Διαγραφή. Της εξής παραγράφου. Result of the entry into force of retroactive provisions of the Acton churches για την παράγραφο λοιπόν αυτή που αναφέρεται στις 300 εκκλησίες που έχασαν το καθεστώ τους. Για την διαγραφή της παραγράφου προτείνει ο συνάδελφος Φρανκ Έγγελ να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα στην 178 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και στη συνέχεια οι 180, 81, 82 είναι ταυτόσιμες. Να περάσουμε στην 184. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 185. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 186. Α, συγγνώμη. 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ. Α, συγγνώμη. Δεν είχε κατατεθεί. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε συνολικά και με ηλεκτρονικό τρόπο το σύνολο της έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δείχνετε κατανόηση γιατί δεν ήταν εξαιρετικά εύκολη η ψηφοφορία. Θα το προσέξετε ως τώρα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ε, ηλεκτρονικά. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ παρακαλώ. Είναι παραπάνω η ψήφη του ΕΛΚ. Σας παρακαλώ φροντίστε το για να είστε όσοι πρέπει. Περισσεύει ακόμα ένα από το ΕΛΚ. Ε, εντάξει, πολύ ωραία. Έναρξη ψηφοφορία παρακαλώ, ηλεκτρονική για το σύνολο του κειμένου. Περά. 31 η ψήφη υπέρ, 19 κατά, 8 εποχέ. Εγκρίθηκε με όλε τι τροπολογίε οι οποίε και ψηφίστηκαν σε αυτή τη μακρά ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την υπομονή σας, για την ε, δουλειά που κάνατε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ίντφελτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο και πριν την ψηφοφορία και θα ήθελα εν συντομία να επανέλθω στο περιστατικό που σημειώθηκε πριν από την ε, ψηφοφορία να δηλώσω για τα πρακτικά ότι διαφωνώ να αφαιρούνται ε, συνθήματα και πλακάτ των βουλευτών, γιατί πολλοί το κάνουν, όσο και να διαφωνώ με το περιεχόμενο τους. Άρα είτε θα πρέπει όλα να απαγορεύονται, είτε όλα να επιτρέπονται. Είτε λοιπόν θεωρώ πραγματικά ότι οι απόψεις που προσπέζεστε είναι ε, απαράδεκτοι, αλλά δεν πιστεύω ότι με το να αφαιρούμε αυτές τις αφήσει και τα διάφορα μηνύματα είναι ο τρόπος να τις ε, καταπολεμήσουμε. Ο πρόεδρος παρατηρεί ότι ε, ε, αυτό ζήτησε να αφαιρεθεί απλά από την οθόνη. Ναι, ζητάτε το λόγο ο εισηγητή. Να μιλήσω λίγο και να κάνω μια παρατήρηση. Δεν είμαι βέβαιο Μίλησα και ευχαρίστησα τις πολιτικές ομάδες και τους εισηγητέ, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και την γραμματεία ασφαλώ τους ε, συμβούλους και τους βοηθούς από όλε τι πολιτικέ ομάδε γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ε, κοπιαστική η δραστηριότητα αυτή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και στα ουγγρικά. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για τη συνεργασία σε μία από τις πιο δύσκολες ψηφοφορίες που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας αυτού του Κοινοβουλίου. Σταματούμε εδώ τις εργασίες μας και θα ξαναρχίσουμε στις 3 ώρα το απόγευμα με την Επίτροπο Ρέντινγκ, υπεύθυνη για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, ε, επανερχόμαστε λοιπόν στις 3 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ.